Meine Κυρίες και κύριοι, δυνάμη του άρθρου 87α 3, η Οικονομική Επιτροπή οθέτησε μία πρόταση ψηφίσματος για τις κατεξουδότητες συνρυθμίσεις της Επιτροπής, για τις τεχνικές κανονιστικές προδιαγραφές, για τις έμεσες συμφωνίες αντιστάθμισης, τις υποχρεώσεις αντιστάθμισης, το Δημόσιο Μητρό, πρόσβαση στις, ε, στους τόπους διαπραγμάτευσης μη χρηματοπιστωτικών ε, αντισυμβαλωμένων, περιορισμό του κινδύνου και έξω χρηματιστικά παράγωγα Πρόκειται για το κείμενο Β700078 του 2013. Προσδιορίζεται η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών στις 12 το μεσημέρι την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου. Ψηφοφορία προβλέπεται για την 5η και έτσι περνώ στην ημερήσια διάταξη με το έκθεση του κυρίου Παπαστάμκου για τα ειδικά μέτρα για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου. Ο κύριος Άτκινς έχει το λόγο όμως για το διαδικαστικό. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να στείλετε ένα μήνυμα προς τον ε, πριν φύγουν ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε από την 1η Τετάρτου ε, προκειμένου να έρθουμε στο Στρασβούργο. Μια και οι γαλλικές αρχές ε, και Air France έχουν ακυρώσει όλες τις πτήσεις από το Charles το αεροδρόμιο του Παρισιού προ το Στρασβούργο. Μήπω θα μπορούσε λοιπόν να κάνετε ένα διάβημα πριν φύγει από το Στρασβούργο με το ιδιωτικό του αεροπλάνο προς τον πρόεδρο τη Γαλλικής Δημοκρατίας. Κύριε Άτκινς, ήσταν ε, συντονιστή στην Επιτροπή για θέματα ε, κανονισμού. Νομίζω ότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτό διαδικαστικό δεν ήταν. Λοιπόν, έχουμε την ψηφοφορία, το κείμενο ολόκληρο καταρχάς ε, και έχουμε την 48 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οι λοιπές τροπολογίες ε, καταπίπτουν ως εκ τούτου και ψηφίζουμε το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα παρακαλώ με μία τροπολογία. Την 49 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και προχωρώ στη ψηφοφορία για το νομοθετικό ψήφισμα. Ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ. έρχεται. Έψηφισαν ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και συγχαρητήρια κύριε Παπαστάμκο. Τώρα έχουμε την έκθεση Μάτο Άντροβερ, ειδικά μέτρα στον τομέα της γεωργίας υπέρ των άκρων απόκεντρων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, α7-321-2011, ε, πρόταση κανονισμού Έχουμε την 115 υπαριθμών τροπολογία συμβαστική. Ποιος μπορεί να την εγκρίνει υπέρ, κατά, άποχες. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίσουμε την πρόταση όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ, κατά. Άποχες. Εγκρίνεται νομοθετικό ψήφισμα. Με μία τροπολογία μετά την πρώτη παράγραφο, 116 τον αριθμό, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα. Ονομαστικά παρακαλώ, άρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε. εγκρίνεται και συγχαρητήρια στον κύριο Μάτο Αντροβέρ. Και τώρα έχουμε την έκθεση του κύριου Ντεμπάκερ, βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, έγγραφο Α7.1 του 2013, με την τροπολογία 34 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα, παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. Και ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστικά παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν οι πάντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Και συγχαρητήρια στον κύριο Ντεμπάκερ. Εύχομαι στους συναδέλφους καλή όρεξη, εφόσον αποχωρούν. Παρακαλώ να αποχωρήσετε ησύχως και ταχαίως, ώστε όσοι θέλετε να αποχωρήσετε, ώστε εκείνοι οι οποίοι θέλουν να παραμείνουν για τις επεξηγήσεις ψήφου να έχουν ησυχία και την προσοχή των συναδέλφων τους. Και τώρα έχουμε τις επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση του κυρίου Παπαστάμκου.